έχουμε 7 ε, ψηφίσματα για το Αζερβαϊτζάν σχετικά με την ελευθερία της ε, έκφρασης και πρώτος ο κύριο Προβέρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, Ευρώπη έχει μια σημαντική εταιρική σχέση και μια πολύ ε, ενθαρρυντική συνεργασία με έξι χώρες Αρμενία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Αζερβαϊτζάν. Η σχέση αυτή βελτιώνει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες αυτές και μπορεί να οδηγήσει σε μια δημοκρατική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αν και σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με την ιστορία της κάθε μίας από αυτές τις χώρες. Πρόκειται για μια ευθύ ε, στρατηγική πολιτική και στα πλαίσια αυτής νομίζω ότι είναι επίγον να συζητηθεί ε, το θέμα των δύο νέων blogger ε, που δικά αυτή τη ενώ υπάρχουν και άλλες ε, τραγικές συνθήκες, όπως η σφαγή 57 ατόμων πρόσφατα που είχαν συγκεντρωθεί για να υποστηρίξουν ε, έναν προεδρικό υποψήφιο στις ε, Φιλιππίνες. Η κατάσταση αυτή στο Αζερβαϊτζάν ε, έχει σχέση με την ε, εταιρική σχέση που έχουμε αναλάβει με τη χώρα αυτή και το ψήφισμα που τίθεται προς πληροφορία σήμερα μπορεί ε, να ε, απευθύνεται όχι μόνο σε μια ε, σκλήρινση της σχέσης του, το, της κυβέρνησης του με την Ευρώπη αλλά μπορεί να αφορά και την τύχη αυτών των δύο νέων και γι' και μπορεί να γίνει πιο δύσκολο, να κάνει πιο δύσκολες τις συνθήκες να αποδοθεί χάρη σε αυτούς τους δύο νέους blogger. Και αυτό ε, κάνει ακόμα πιο σοβαρό το γεγονός ότι σήμερα δεχτήκαμε να μην συζητήσουμε την υπόθεση Χάινταρ για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή της. Μου φαίνεται ότι είναι αντιφατικό στην ίδια ε, συνεδρίαση να ε, τεθούν ε, σε ψηφοφορία δύο ψηφίσματα εντελώς διαφορετικού ύφους, ένα για τη Λευκορωσία και ένα για το Αζερβαϊτζάν Αζερβαϊτζάν ε, όταν ε, έχουν ε, τόσο μεγάλη σημασία αυτές οι δύο χώρες για την ανατολική εταιρική μας σχέση. Για ένα λεπτό, συντάκτρια Κέριγκα Τσου Όντενμπεργκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στι 11 Νοεμβρίου, όταν γιορτάζαμε τον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, στην, στο Αζερβαϊτζάν, καταδικάστηκαν δημοσιογράφοι σε ποινές ε, πολιτούς φυλάκισης ε, διότι είχαν ε, κατηγορήσει για τη διαφθορά την κυβέρνηση και τις αρχές. Το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα χωρίς ελευθερίες και ελευθερία του τύπου και είναι η 146η έκτη χώρα από 175 χώρες όσον αφορά την ελευθερία του εκφράζεστε. Είναι πολύ ανησυχητικά τα στοιχεία τα οποία ε, παίρνουμε από τις ε, μονάδες ε, και τις, τους όσους αναφέρουν τα όσα συμβαίνουν στο Αζερβαϊτζάν. Και σε σχέση με τις αρχές και την έλλειψη των ε, αδειών ε, που δεν δίνουν για ε, αλλοδαπούς δημοσιογράφους να μπορέσουν να πούν το τι συμβαίνει στο ίδιο το Αζερμπαϊζάν. Πρέπει επίσης να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να αρχίσει να ασκείται μεγαλύτερη πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη χώρα και να ασκηθεί πίεση να ελευθερωθούν οι δημοσιογράφοι και να αναθεωρηθούν τα νομικά αυτά πλαίσια. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκέριγκερ Ντεόντενμπεργκ και τώρα στη συνέχεια πάλι ο συντάκτρια κυρία Σάκε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και αγαπητοί συνάδελφοι. Το Αζερβαϊτζάν έχει υπογράψει διάφορες εταιρικέ σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενεργοποιείται στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, καθώς επίσης και τη Ανατολική Εταιρική Σχέση, που δεν σχετίζονται μόνο με το εμπόριο. Το Αζερβαϊτζάν έχει υπογράψει την δέσμευση να σέβεται τη δημοκρατία ε, και το κράτος δικαίου. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά απειλούνται από το σημερινό καθεστώς του Αζερβαϊτζάν. Σήμερα τονίζουμε την περίπτωση του Εμίν Μιλή και του Αδνάν Χάτζι Τζάντε, ε, που ε, είναι ε, εκφραστές μιας κατάστασης στην ελευθερία της έκφρασης που πάει πολύ βαθύτερα από την δική τους ατομική περίπτωση. Ε, το γεγονός είναι ότι δεν ξέρουμε ε, ούτε καν γιατί βρίσκονται στη φυλακή, γιατί δεν έχουν γίνει δεκτά διάφορα αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη τους και φαίνεται με τα διεθνή κριτήρια ότι είναι κατασκευασμένα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου. Ε, το Αζερβαϊτζάν πρέπει να ε, σεβαστεί όλες τις ε, δεσμεύσεις και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί το Αζερβαϊτζάν αξιόπιστο εταίρο ούτε και στις εμπορικές σχέσεις. Το ψήφισμα αυτό καλεί την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να αρχίσει να νομιμοποιεί τη θέση της στην διεθνή κοινότητα ξεκινώντας από το σεβασμό προς τους πολίτες της χώρας και ε, σεβόμενοι το κράτος δικαίου. Χθες δώσαμε το βραβείο Ζαχάροφ και ε, ακούσαμε ένα πολύ εντυπωσιακό λόγο από τον κύριο Κόβαλοφ ε, που είπε ότι ο φόβος αντιμετωπίζεται μόνο με την ελευθερία σκέψης και η ελευθερία σκέψης μπορεί να εκφραστεί μόνο όταν εξασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης και όταν μπορούμε ε, να ακούμε ε, τέτοιους ανθρώπους που απλώς εκφράζουν ε, την αντιπολίτευση προς την κυβέρνησή τους. Αυτό εμείς πρέπει να το εγγυηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους μέσα από όλες τις εταιρικέ σχέσεις που έχουμε με το Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφε Σάκε. Στη συνέχεια πάλι ο συντάκτρια η κυρία Λούνα Τσέκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ήδη οι πρόεδροι σας ανέφεραν κάποια στοιχεία από αυτό το ψήφισμα. Πρόκειται εδώ κυρίω αίτιο για αυτή τη σύνταξη αυτού του ψηφίσματο ήταν κάτι από τον Ιούλιο 2009. Δύο νέοι μπλόκερ, οι Μίλη και Χατζή Ζαντε, συνελήφθησαν μια και είχαν και προηγούμενα υποστεί επίθεση σε ένα εστιατόριο. Μετά του πήγαν σε ένα αστυνομικό σταθμό όπου έγιναν καταγγελίε Μετά ε, ξεκίνησε μια δίκη εις βάρος τους, μια διαδικασία δικαστική που όλους τους διεθνούς, διεθνείς παρατηρητές στην Amnesty International και σε όλους τους άλλους ε, θεωρήθηκε ως μη δίκαιη δίκη για παράδειγμα, σε σχέση με το βίντεο σε εκείνο το εστιατόριο που απαθανατίστηκε, απαθανάτησε εκείνες τις στιγμές και έδειξε ότι δεν ήταν αυτοί οι δύο νέοι blogger, αλλά άλλοι οι οποίοι είχαν ε, συμμετάσχει σε βιοπραγίες. Πρόκειται εδώ για κάτι λοιπόν, για μια διαδικασία, μια δίκη που δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ενός κράτους δικαίου. Και ελπίζω ότι όταν θα γίνει αυτή η δίκη, όλα θα πρέπει να αποκαλυφθούν και να διχθούν όπως, όπως έγιναν. Χαίρομαι γιατί καταλήξαμε σε μια πρόταση ψηφίσματος από σχεδόν όλες τι κοινοβουλευτικές ομάδες. Λυπούμε που η κοινοβουλευτική ομάδα του συναδέφου Προβέρα δεν ακολούθησε τη δική μας ε, γραμμή, τη δική μας πορεία. Και ότι θα πρέπει τώρα να επιληθεί το θέμα αυτό με τις διπλωματικές διαδικασίες κτλ. Θα έλεγα όμως κύριε Προβέρα ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σε εταιρική σχέση βρίσκεται με το Κοινοβούλιο του Αζερβαϊτζάν πρέπει να τοποθετηθεί με σαφήνεια γι' αυτό. Τα, τα θεμέλια μας είναι τα, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν είναι αναγκαίο να εκφραζόμαστε υπέρ αυτών και για την πνευματική ελευθερία και την ελευθερία του εκφράζεστε παντού στον κόσμο. Ο πρόεδρο Αλίεφ του Αζερβαϊτζάν ο ίδιο το έχει πει πολύ συχνά, πολλέ φορέ πόσο σημαντικά είναι τα δικαιώματα αυτά και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Είναι λοιπόν δική μα δουλειά να υπενθυμίζουμε αυτό το πράγμα ξανά και πάλι. Και έτσι με αυτή την πρόταση ψηφίσματος θέλουμε και μέσω τη εταιρική σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου του Αζερβαϊτζάν και Ευρωκοινοβουλίου να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ συνάδελφε Λούνατσεκ. Στη συνέχεια πάλι ο συντάκτη, ο κύριο Higgins παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Εκτός, εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Yes, it is on, Εδώ είναι, λέει ο μιλητής. Καλωσορίζω την προσοχή που δίδεται στις φρικτέ και μόνιμες παραβιάσει των δικαιωμάτων των ανθρώπων στο Ατζερμπαϊτζάν. Δεν υπάρχει ελευθεροτυπία, ε, δεκάδε δημοσιογράφοι φυλακίζονται, κάποιοι σκοτώνονται τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ζητήσουμε κατά πόσον το καθεστώς, γιατί το καθεστώ Αλίεφ εφαρμόζει τέτοια βία, προσπαθώντας προφανώς να καλύψει το καθεστώς της τεράστιας διαφθοράς που υπάρχει στην χώρα αυτή. Η κυρίαρχη ελίτ έχει πλουτίσει απίθανα χάρη κυρίως στη βιομηχανία του φυσικού αερίου και του, πετρελαίου. Ωστόσο, το 90% του πληθυσμού του Αζερβαϊτζάν ζουν υπό συνθήκε τέλεια φτώχεια και δεν έχουν κερδίσει τίποτα από του τεράστιου πόρου τη χώρα. Βεβαίω, η κυβέρνηση και οι πολυεθνικές λειτουργούν με υποκρισία. Ε, τα βρίσκουν με τον καθεστώς, ευκολύνουν έτσι τις δουλειές τους και Προφανώς οι επιχειρήσεις μαζικά, αποκτούν μαζικά κέρδη από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων που ανήκουν στο λαό του Αζερβαϊτζάν. Οι υπόλοιπε κυβερνήσει λοιπόν θα έπρεπε να πούν γιατί δεν ζητούν ε, να χρησιμοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθεί το πετρέλαιο για τη βελτίωση της, ε, των συνδικών ζωής του λαού. Το Κοινοβούλιο παρουσίασαν σωστά την ε, σκληρή καταδίκη τους ε, από την απαγόρευση, στην απαγόρευση της ελευθερίας έκφρασης των θέσεων στο Αζερβαϊτζάν. Αλλά θα έπρεπε ταυτόχρονα να καταδικάσουμε και την ε, καταπιεστική καταστολή των διαδηλωτών από την δανική αστυνομία στην Κοπενχάγη όπου χιλιάδες Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωναν ειρηνικά, ωστόσο συνελήφθηκαν, ε, τους πέρασαν χειροπέδες και τους άφησαν επί ώρες να περιμένουν στο κρύο. Απλά και μόνο ε, συνάδελφοι δικοί μας τέθηκαν σε προληπτική ε, σύλληψη. Αυτό που ισχύει για το Αζερμπαϊτζάν θα έπρεπε να ισχύει και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Higgins. Ως συντάκτης ακολουθεί ο κύριος Λεγκούτκο. Κύριε Πρόεδρε, στο Αζερβαϊτζάν, αν κάποιος επικρίνει την κυβέρνηση και με ευγενικά λόγια ακόμα, φυλακίζεσαι. Δύο άτομα φυλακίστηκαν και, με, με μεγάλες ποινές. Τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει σωστό σύστημα απονομής δικαίου στη χώρα και δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Πρόκειται για ένα αυταρχικό σύστημα το οποίο θέλει να επεκταθεί και πλήττει όσους είναι αντίθετοι με αυτό. Εμείς τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα θα έπρεπε να παρέμβουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αδικίες. Αυτό το κάνουμε και τώρα. Μερικές φορές η δράση μας είναι αποτελεσματική. Ωστόσο είναι πολύ πιο δύσκολο να ζητήσουμε για θεσμικές αλλαγές στη χώρα Μέχρι τώρα οι προσπάθειές μας δεν ήταν επιτυχεί στον τομέα αυτό. Εν μέρη, διότι μερικές φορές έχουμε δείχνουμε μεγαλύτερη κατανόηση σε ορισμένου τυράννου και λιγότερη σε άλλου. Ακούσαμε σήμερα τους χτες τους εκπροσώπους του Memorial να μιλούν για την κατάσταση εκεί σε πολλές ευκαιρίες. Επίσης, Υπάρχουν προβλήματα διότι εν μέρη η διαδικασία της μεταβολής από ένα αυταρχικό σε ένα δημοκρατικό καθεστώς είναι δύσκολη. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία που απαιτεί χρόνο, πολύ χρόνο. Δυστυχώς το συμπέρασμα είναι απεσιόδοξο, ωστόσο πιστεύω ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να επιμείνουμε ασκώντας πίεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε Λεγκούρκο. Τελευταίο ε, από βράσεων συντακτών, ο κύριο Κέλαμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή αυτή τη χρονιά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μια δήλωση για την ελευθερία των μέσων και του τύπου στο Αζερβαϊτζάν και μάλιστα αφού είχε εκφραστεί η ανησυχία για την ελευθερία του τύπου στην τακτική συνεδρίαση με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Αζερβαϊτζάν λυπούμε που δεν υπήρξε feedback, κάποια αντίδραση. Γι' αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στεναρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι το τελευταίο ψήφισμα αυτό το οποίο θα εγκρίνουμε φέτος το 2009. Το κύριο μέλημα της ομάδας ε, του ΕΛΚ και χαίρομαι για το ότι όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες συμμερίζονται αυτό το μέλημα είναι η επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων του τύπου σε αυτή τη χώρα. Η διαδεδομένη μέθοδος ε, ε, του εκφοβισμού, των, της καταστολής και των διώξεων, πράγμα το οποίο είναι φρικτό. Ζητούμε από τις αρχές του Αζερβαϊτζάν να απελευθερώσουν τους δημοσιογράφους που έχουν φυλακιστεί άμεσα. Αυτό αφορά και τους νεαρούς bloggers. Τώρα, το δεύτερο είναι μια πρόσφατη απόφαση των αρχών του Αζερβαϊτζάν να άρουν την άδεια λειτουργίας του ραδιοσταθμού FM και σε σχέση και με άλλους ε, ραδιοσταθμούς όπως ε, το BBC, το ε, Radio Free Europe, Radio Liberty λοιπά Οι ανεξάρτητες πηγές και φωνές της ενημέρωσης εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θέλω να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι για την παράγραφο 7 σε μια προφορική τροποποίηση. Όχι μόνο να εκφράσουμε την θλίψη μας για αυτή την κατάσταση, αλλά να απευθύνουμε κατεπηγόντως έκκληση στην κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν να άρει αυτή την απόφαση και να ανανεώσει την άδεια λειτουργίας αυτού του σταθμού, ραδιοφωνικού σταθμού. Το ε, δικαίωμα στην ελευθερία του εκφράζεστε είναι κλειδί για την κοινωνία των πολιτών, όπως μας είπε ο Σεργέη Καβαλιόφ στο ε, σώμα εχθές. Αυτό ε, εφαρμόζεται πλήρως και ισχύει για τις σχέσεις μας με το Αζερμπαϊτζάν και αυτό πρέπει να τους πούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλαμ και ακολουθούν τώρα οι αγορητές εξ των πολιτικών ομάδων η κυρία Αντρικιένε. Ένα λεπτό για την ομάδα του ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Αζερβαϊτζάν είναι ένα μεγάλο, μεγάλο τμήμα της ε, ε, ε, μεγάλος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρος ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικό είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεν είναι τα πάντα. Το Αζερμπαϊτζάν έχει δεσμευτεί να δουλέψει και να αγωνιστεί για μια δημοκρατική πλουραλιστική κοινωνία, όπω απαιτεί η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία, καλά και η ε, πολιτική ε, συνεργασία στην Ανατολή, στην οποία θέλει να μετάσχει το Αζερμπαϊτζάν θέλει, πρέπει να ε, υποστηρίξουμε τα θετικά βήματα του Πρόεδρου να απελευθερώσει για παράδειγμα 119 φυλακισμένους με, το, με, το, πολλούς ε, ωστόσο, η κατάσταση των μέσων ενημέρωσης επιδεινώνεται. Υπάρχουν περιπτώσεις που το αποδεικνύουν αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά τις άδειες ε, λειτουργίες του BBC ή του Radio Free Europe. Δεν θα πρέπει να γνωρίσουμε την κατάσταση. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στο Αζερβαϊτζάν ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα να μιλά ελεύθερα, έστω και αν επικρίνει την κυβέρνηση. Τελειώνω. Αυτό είναι η βασική αρχή μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Και το δημοκρατικό Αζερβαϊτζάν πρέπει να είναι διακόπτεται η ομιλήτρια. Σα ευχαριστούμε συνάδελφε καινέ. Ναι. Για ένα λεπτό στη συνέχεια εξ ονόματο τη ΕΣΕΜΠΕ κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η ελευθερία ε, έκφραση είναι βάση της δημοκρατίας. Το Αζερβαϊτζάν επικύρωσε τη σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και δεσμεύτηκε και δεσμεύτηκε να τηρεί τα δικαιώματα αυτά. Πρέπει ο κόσμος να μπορεί να εκφράσει τις θέσεις του και να μην ενοχλείται από την, από την κυβέρνηση. Το Αζερβαϊτζάν δεσμεύτηκε να μην ε, παραβιάζει τα δικαιώματα του ανθρώπου και να υλοποιεί τι αρχές της εταιρική σχέσης προς την Ανατολή που, συν, που συμφωνήσαμε. Τα τελευταίο καιρό ωστόσο απειλείται το δικαίωμα έκφρασης ε, στο Αζερβαϊτζάν αλλά και το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Ε, χρησιμοποιούνται μέσα παρεμπόδιση ε, των εργασιών και, ενώ, και των δημοσιογράφων. Ζητούμε από το Αζερβαϊτζάν να βελτιώσει το σύστημα προστασία των δικαιωμάτων ανθρώπων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε συνάδελφε Μπλίνκεβιτσιούτε. Στη συνέχεια, εξ ονόματο τη ομάδα HCR, ο συνάδελφο Τσαρνέτσκι, δύο λεπτά παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Για άλλη μια φορά, το Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν εγγράφεται στην ημερήσια διάταξή μα Να σα υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη φοιτεία μα εγκρίναμε τρία ψηφίσματα που αφορούσαν το Αζερβαϊτζάν για την ελευθερία του τύπου, Μεταξύ αυτών κάναμε λόγο επίσης και για τον Νότιο Κάφκασο συμπεριλαμβανομένου και του Αζερμπαϊτζάν. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν για αυτή τη χώρα και θέλουμε να πάει καλά και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Είναι μια χώρα που προσπαθεί να βρει την πορεία της και βήμα προς βήμα όλο και πιο κοντά φτάνει προς τον δυτικό κόσμο και τον προσεγγίζει και παρεκκλίνει και απέχει περισσότερο από την Ανατολή πλέον και αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμάμε και με θετικό ενδιαφέρον στρεφόμαστε προς αυτή τη χώρα και τις αρχές της όμως οι καλές προθέσεις μας και η ε, καλή αυτή στάση δεν μπορεί να δεχθεί να επιβάλλονται κάποια πράγματα να αποφύγουμε να μην μιλάμε για παράδειγμα για πράγματα όπως όταν συλλαμβάνονται και φυλακίζονται bloggers Γι' αυτό λοιπόν επειδή ακριβώς εξέφρασαν τις απόψεις τους ε, για τους κρατούντες και την ίδια την κυβέρνηση και φυλακίστηκαν. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Αζερβαϊτζάν, διότι διεξάγεται μια πολιτική συζήτηση σε αυτήν τη χώρα αν θα πρέπει να προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρώπη ή την Ρωσία. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλους εκείνους που επιθυμούν να προσεγγίσουν τον δυτικό κόσμο. Υποστηρίζοντάς τους όμως πρέπει να ασκήσουμε και πίεση ταυτόχρονα για να είναι σεβαστές οι σημαντικές αξίες, δηλαδή η ελευθερία, η ελευθερία του εκφράζεστε, η ελευθερία του τύπου, αυτές οι θεμελιώδεις αξίες και αρχές. Είμαι, ε, πιστεύω ότι το Αζερβαϊτζάν αντιμετωπίζει σήμερα μια δύσκολη κατάσταση, επειδή προσπαθεί η Ρωσία να επανασυγκροτήσει την σφαίρα επιρροής της και, να και υποστηρίζοντας τις αρχές του Αζερβαϊτζάν πρέπει να τους πούμε όμως ότι δεν ακολουθούν τη σωστή πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τη, στη συνέχεια θα λάβει τώρα τον λόγο για την ομάδα της ΕΦΤΣΕ ο συνάδελφος Φάσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ελευθεροτυπία είναι βασική διάσταση μιας δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, παρακολούθησε τις δραστηριότητε που είχαν στόχο ε, να αμφισβητήσουν τις, ε, την αμφίβολη συμπεριφορά κάποιων κυβερνητικών αξιωματούχων στο Αζερμπαϊτζάν. Θέλω να εκφράσω λοιπόν τις ανησυχίες μου για τις συνέπειες των αστυνομικών διώξεων κατά νέων ανθρώπων που απλά ε, θέλουν να δείξουν και να αναδείξουν τα προβλήματα της χώρας τους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κάποιες απαράδεκτες δηλώσεις που προέρχονται από το Αζερβαϊτζάν. Είμαι ε, Προφανώ είναι κρίσιμη η κατάσταση του Αζερβαϊτζάν, αλλά ε, δεν θα έπρεπε να γνωρούμε ότι ε, το Κοινοβούλιο είχε πολύ επιθετικές, ε, είχε μια πολύ επιθετική στάση στις Φιλιππίνες, όπου 57 άτομα δολοφονήθηκαν. Την ίδια προσοχή πρέπει να τη δίνουμε και παντού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Βαντερστού που δεν είναι παρόν για τους μη εγγεγραμμένους, Για να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Πόσολ δύο λεπτά. Εκτός... Κύριε Πρόεδρε, στις πρώτες ευρωεκλογές ε, είχα την ε, τιμή να συνδράμω και εγώ σε αυτή την ε, στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρώπης. Το 1994 είχα την τιμή με τον συνάδελφο Σούλτς να συνεχίσω αυτή την ε, στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την οποία είμαστε περήφανοι και γι' αυτό με σόκαρ το γεγονό ότι ο συνάδελφο Προβέρα απευθύνθηκε έτσι για τον κύριο Σούλτ, το, ο οποίος δεν το άξιζε και μίλησε για τις απειλές ε, του καθεστώτος ε, του Αζερβαϊτζάν κατά των ατόμων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλήσαμε για το, το βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θυμάμαι ότι όταν ε, ταχθήκαμε υπέρ του Ζαχάροφ, του Λανσμπέργκης, είχαμε πει ότι σας παρακαλώ ας μην προκαλέσουμε ζημιές, ας αφήσουμε να δράσει η διπλωματική οδός. Σήμερα είναι σαφές ότι το Ευρωκοινοβούλιο ύψωσε τον άστημά τους. Γι' αυτά λοιπόν ας συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. Ας αφήσουμε τα πράγματα αυτά που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την κομματική πολιτική. Είπαν οι συνάδελφοι στην προηγούμενη ελλομέλεια, ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Κίνα. Σήμερα υπήρξε ένα άλλο θέμα, η Δυτική Σαχάρα. Ίσως να είναι δικαιολογημένα όλα αυτά, αλλά ειλικρινά αναρωτιέμαι για την ποιότητα του έργου μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση του Αζερμπάιτζαν γιατί είναι μακρά η ιστορία της χώρας αυτής και τώρα πια σήμερα ξεκινά αργά και οδυνηρά ο εκδημοκρατισμό τη χώρα. Λοιπόν, σε αυτό το δρόμο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ, συνάδελφε, να Ένα λεπτό, κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή. Θα πρέπει να φροντίσουμε το Αζερβαϊτζάν να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και θα πρέπει να απελευθερωθούν και οι δύο νέοι αυτοί που κρατούνται. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά αποδεκτικά στοιχεία και όλα αυτά θα πρέπει να συμβούν κατεπηγόντω γιατί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία στη χώρα αυτή έχει επιδεινωθεί δραματικά. Αυτό το καταδεικνύουν και οι τελευταίες εκθέσεις του ΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτεί για την ελευθεροτυπία, θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, γιατί μεσοκάρτο σοκάρει το γεγονός και η διαδικασία που ακολουθήσαμε σήμερα σε ό,τι αφορά την κυρία Χάινταρ. Γιατί η καλή συνεργασία μεταξύ Μαροκινών και Ισπανικών αρχών θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στην επίλυση του θέματος, του δράματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Στη διαδικασία Catch the Eye, ένα λεπτό ο συνάδελφος Τσβίφκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω το άρθρο 47 του συντάγματος του Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή όλοι έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας σκέψης και λόγου. Όμως αυτά είναι κενά λόγια. Δεν τηρείται το Σύνταγμα. Για πέντε χρόνια υπήρξα μέλος της αντιπροσωπείας συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Νοτιού Καυκάσου. Έχω επισκεφθεί το Αζερμπαϊτζάν ε, στο πλαίσιο της κοινή κοινοβουλευτική ε, συνέλευσης και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι με προκατασκευασμένες κατηγορίες στέλνονται στη φυλακή και όταν αρρωστήσουν δεν λαμβάνουν ε, ιατρική βοήθεια. Είχαμε μάλιστα και ένα μοιραίο περιστατικό, ένας ε, δημοσιογράφος ο οποίος κατέληξε διότι δεν του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Έχω επισκεφθεί φυλακές στο Αζερμπαϊτζάν πρέπει να σας πω ότι τα πρότυπα, οι συνθήκες απέχουν μακράν αυτών που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε ότι το Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να τηρεί το σύνταγμά του. Ευχαριστώ. Δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Επίτροπο Σαμέσκι. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, το Αζερβαϊτζάν είναι σημαντικό, σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω παραγωγό χώρα και ω χώρα διέλευση. Αλλά είναι σημαντική για την περιφερειακή σταθερότητα του Καυκάσου. Είναι μία από τι έξι χώρε τη Ανατολική Εταιρική Σχέση. Δίνουμε μεγάλη σημασία στον σεβασμό των κοινών αξιών και τη βελτίωση των σχέσεων. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία ισχύει εδώ και 10 χρόνια. Ωστόσο, το Αζερβαϊτζάν εξέφρασε το ενδιαφέρον του να έχει ακόμα στενότερε σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάπτοντα μια συμφωνία σύνδεση για αντικατάσταση της πρώτη συμφωνίας. Με την απόφαση το Σεπτέμβριο της Ευρω... της... του Υπουργών, των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μια τέτοιας συμφωνίας με τις χώρες του Νοτιού Καυκάσου, οι συζητήσει για τη ε, διαδικασία αυτή συνεχίζονται με το Αζερβαϊτζάν. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, το καθεστώ των διαπραγματεύσεων με κάθε χώρα του Νοτιού Καυκάσου θα είναι υπό την αίρεση τη στήριξη των, ανα... των ε, απαραίτητων ε, προϋποθέσεων, σεβασμό του κράτους δικαίου, ε, δικαιώματα ελευθερίες, αρχές ελεύθερης οικονομίας και βιώσιμη διακυβέρνηση. Κάθε χρόνο κάνουμε μια αξιολόγηση και καταγράφουμε την πρόοδο που κάθε χώρα εταίρος πέτυχε για την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσεως βάσει της πολιτικής μας. Ξεκινήσαμε την προπαρασκευαστική δραστηριότητα για την έκθεση για το 2009. Δεν θέλω να προδικάσω την έκθεσή μας, θέλω να κάνω ωστόσο κάποιες παρατηρήσεις, ιδίω ως προς την κατάσταση που αφορά τις ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην έκθεση για το 2008 αναφέραμε και παραθέτω ότι το Αζερβαϊτζάν προόδευσε αρκετά στην, ε, στον τομέα αυτό, αλλά δεν έχει πολύ, πολύ σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Έκτοτε, δυστυχώ, είχαμε αρνητικέ εξελίξεις. Φερρυπίν, συνταγματική αλλαγή, κατάργηση του ορίου επανεκλογής του αρχηγού του κράτους, κράτηση και καταδίκη δύο μπλόγκερ. Άλλε αρνητικέ εξελίξεις περιλαμβάνουν επίσης την συνέχιση των διώξεων των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των, των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και των δημοσιογράφων, πέραν της επιπλέον, των, των επιπλέον περιορισμών στην ελευθεροτυπία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα επίπεδα ανέφερε τα ζητήματα αυτά στις αρχές και θα συνεχίσει να το κάνει. Ταυτόχρονα η Επιτροπή κινητοποιεί μια σειρά εργαλείων για να βοηθήσει τη χώρα αυτή για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται με τη νέα συμφωνία. Χρησιμοποιούμε τη συμφωνία μέσω του εργαλείου ε, πολιτικής γειτονίας. Δίνουμε στοχοθετημένη υποστήριξη σε ένα ε, σφαιρικό σύστημα ενίσχυσης των θεσμών με σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνουν ε, διαστάσεις κράτους δικαίου και ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος. Το επίσης το Αζερβαϊτζάν θα τύχει βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την ε, Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Με την υφιστάμενη συμφωνία προτείνουμε εν τέλος, τέλος να δημιουργήσουμε μια επιτροπή που θα ενισχύει τους τομείς δικαιοσύνης, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που θα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Επιτροπέ Σαμίσκι, Να περάσουμε τώρα στις ε, ψηφοφορίες για έξι ψηφίσματα για την ομοφιλοφιλία. Καταρχάς, να κοιτάξουμε το κοινό ψήφισμα έξι ομάδων που θα αντικαταστήσουν τα ψηφίσματα αυτά. Να ψηφίσουμε λοιπόν την παράγραφο 6 του αρχικού κειμένου.